Καλημέρα. Καθίστε παρακαλώ. Είμαστε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Καλωσορίζω εδώ τον κύριο Hans Χόχερφόρστ, που είναι πρόεδρος του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, και τον κύριο Λίκάνεν, που είναι ο πρόεδρος του, των τραστής του Ιδρύματος Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ιδιωτικό οργανισμό που ασχολείται με τα λογιστικά πρότυπα. Θα ενσωματωθεί μάλιστα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω μιας ε, διαδικασίας έγκρισης. Ο κύριος Χόχερ είχε διάφορες θέσεις στην Ολλανδική κυβέρνηση, ήταν υπουργό Οικονομικών και ο κύριος Λικάνεν ήταν δύο φορές διοικητής της Τράπεζας της Φιλανδίας. Όπως επίσης και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επίτροπος και υπουργό Οικονομικών στην Ολλανδία από το 1987 μέχρι το 2009. Συνεπώς, θα δώσω το λόγο στον κύριο Χόχερφορστ για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα κάποια ιστορικά δεδομένα. Ο Πολ Βόλκερ που ήταν ε, διοικητής της ΦΕΤ, απεβίωσε και ήταν ένας από τους ε, αξιωματούχους που εκτιμούσαμε περισσότερο. Εγώ ήμουνα ο πρώτος πρόεδρος ε, των τραστής του IFRS. Και όταν εκείνος είχε μιλήσει για το κόσμο μετά την κατάρρευση Λίμαν και τα λοιπά, είχε πει ότι έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή στην αναφορά προτύπων. Διαφάνεια παγκοσμίω. Τότε ακριβώς ήταν που και η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να εγκρίνει διεθνή λογιστικά πρότυπα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο. Γιατί αυτό γινόταν με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Αυτά βέβαια ήταν πριν από 18 χρόνια. Έτσι. Πολλά έγιναν από τότε, αλλά τότε ξεκινήσαμε. Η δομή τώρα, η διάρθρωση έχει αλλάξει. Γιατί σήμερα έχουμε και το ελεγκτικό συμβούλιο που αποτελείται από αρχές που προστατεύει ε, τα συμφέροντα του κοινού και μάλιστα αυτή τη βδομάδα θα συναντηθούμε εδώ στις Βρυξέλλες. Πάντως η Τραστής είναι το σώμα το οποίο εγώ προεδρεύω και εγώ εδώ ε, μιλάω ε, για κάποια πράγματα και ο κύριος Χόκαρφος θα μιλήσει για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους ε, τραστείς. Ποιος είναι ο ρόλος τους. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εξετάζουν τα στατιστικά ζητήματα που καταλήγουν σε διεθνή λογιστικά πρότυπα και εξετάζουμε το περιεχόμενο. Δεύτερον, θέλουμε να κοιτάμε και τους ικανονικούς διακανονισμούς και να εγκρίνουμε τον ετήσιο προπολογισμό. Τρίτον, είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ορίζουμε τα μέλη του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τον Πρόεδρο. Οι τραστείς δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Και τέλος, στόχος μας είναι να κοιτάμε και τις λειτουργικές διαδικασίες με διαφάνεια, γιατί αυτό καθορίζει το έργο μας. Η διαφάνεια, όταν τα πρότυπα γίνονται αποδεκτά παγκοσμίω, είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους. Ε, για την εμπιστοσύνη, για το κοινό, για τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό τι διαδικασία ακολουθούμε και πρέπει να ξέρουν πώς καταλήξαμε σε αυτά τα πρότυπα. Οπότε θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο και μετά ευχαρίστω να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ πολύ εκεί. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων που με κάλεσαν εδώ πάλι. Έχω έρθει τουλάχιστον 10 φορές εδώ και να πάλι. Όπως είπε και ο Ελκή, ξεκινήσαμε πριν από 18-19 χρόνια και έκτοτε πάνω από 140 χώρες έχουν υιοθετήσει τα πρότυπά μας. Και αυτό είναι κάτι εκπληκτικό. Γιατί έχουμε καταλήξει να είμαστε από το πιο σημαντικό σώμα διεθνώς και τα πρότυπά μας ε, συνεχώς τηρούνται και παρά τις τάσεις παγκοσμιοποίησης και τα λοιπά, είναι τα δικά μας πρότυπα τα οποία προέχουν. Οι επενδυτές από την άλλη μεριά κατανοούν και εμπιστεύονται έτσι τις οικονομικές δηλώσεις από που και αν έρχονται, των συνταξιδοτικών ταμείων για παράδειγμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας ακριβώς να υπάρχουν σωστές, καλές ε, πληροφορίες χρηματοπιστωτικές. Είναι σημαντικό και για τις πολυεθνικές να χρησιμοποιούν την ίδια λογιστική γλώσσα όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή. Είναι δημόσιο αγαθό. Βέβαια υπάρχει κάποια εξαίρεση όπου ακόμα δεν υπάρχουν ε, παγκόσμια λογιστικά πρότυπα. Και ήθελα ακριβώς για αυτή την εξαίρεση να σας μιλήσω. Και πρόκειται ακριβώς για το πρότυπο IFRS 17. Πρόκειται για τα ασφαλιστικά συμβόλαια που πρέπει ακόμα να περάσουν και εκεί τα πρότυπα αυτά. Και έρχομαι στην επόμενη διαφάνεια. Υπάρχει τώρα μία ποικιλομορφία λογιστικών ε, προτύπων στα ασφαλιστικά ανά τον κόσμο και τα περισσότερα από αυτά είναι ξεπερασμένα. Χρησιμοποιείται το κόστος και το όφελος, ε, δηλαδή ε, τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώνουν οι άνθρωποι επιχειρήσεις για μια ασφάλεια ζωής ας πούμε. Και τα επιτόκια έχουν πέσει φοβερά τα τελευταία 10-20 χρόνια. Τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγκάζονται να αγοράσουν κυβερνητικά ομόλογα, τα οποία έχουν μερικές φορές και αρνητικές αποδόσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων αποτελεί μια τεράστια δυσκολία για τις ασφαλιστικές εταιρείες και γίνονται πολλά λογιστικά ανά τον κόσμο που δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα. Δεν αντικατοπτρίζουν αυτά τα χαμηλά επιτόκια. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή το δικό μας το Συμβούλιο προσπαθεί λοιπόν να ε, συμπεριλάβει και αυτά τα πρότυπα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ίσως λοιπόν μπορώ επίσης στην επόμενη διαφάνεια να σας δείξω κάτι ακόμα. Η διαφάνεια αυτή δείχνει τις διαφορές ανάμεσα ε, στις εγγυήσεις που έχουν προσφέρει στους πελάτες τους ασφαλιστικές εταιρείες και τις αποδόσεις που έχουν πετύχει από τα κυβερνητικό ομόλογα και βλέπετε ότι έχουμε αρνητικά στοιχεία. Κορέα, Ιαπωνία, ε, Ταϊβάν, ε, μέρος της γερμανικής αγοράς, εκεί οι ασφαλιστές βρίσκονται από κάτω. αρνητικό έχουν αρνητική απόδοση στις ε, επενδύσεις τους. Αυτό λοιπόν δείχνει το πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό δεν θα ήταν τόσο σοβαρό εάν τα λογιστικά πρότυπα ήταν τα σωστά από την αρχή. Αν προσαρμόζονταν δηλαδή στα επιτόκια ε, της κάθε στιγμής και δεν βασιζόντουσαν στα ιστορικά επιτόκια που ίσχυαν κάποτε και που δεν ισχύουν πια. Άρα λοιπόν είναι καλό παράδειγμα για να καταλάβει κανείς πώς μπορούν να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις αν υπάρχουν σωστά λογιστικά πρότυπα. Επόμενη διαφάνεια. <clears throat> Έχουμε λοιπόν το πρότυπο αυτό 17 δεν θέλω να μπω εδώ σε λεπτομέρειες, είναι βέβαια ιδιαίτερα περίπλοκη η περίπτωση αυτού του προτύπου και της έγκρισής του, πάντως δεν βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα, βασίζεται σε σημερινά δεδομένα και σημερινές υποθέσεις ώστε να αντικατοπτρίσουν τα πρότυπα αυτά το πραγματικό κόστος των επιλογών και των εγγύσεων. Και επίσης η αναγνώριση ε, του, των εσόδων επίσης αναγνωρίζεται, γιατί πολλές ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρίζουν και τις αποταμιεύσεις των ε, αποταμιευτών. Το IFRS 17 δείχνει επίσης πόσο καλή είναι η συνεργασία μας με την Ευρώπη για να έχουμε τα πρότυπα αυτά. Είμαστε μια μικρή ομάδα ανθρώπων στο Λονδίνο και χρειαζόμαστε πραγματογνωμοσύνη από τον έξω κόσμο για να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Έχουμε λοιπόν ε, διαδικασία ε, βάσει της οποίας ε, ακούμε πολύ κόσμο. Και στο στάδιο υλοποίηση του προτύπου, που συνήθως είναι περίπλοκη, πολλά θέματα ετέθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον κόσμο. Ρωτάνε, θα μπορούσε η υλοποίηση να γίνει πιο απλή, να υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, στο πρότυπο, για παράδειγμα. Και εδώ βλέπετε <coughs> από τα 10 θέματα, τα 6 έρχονται από το ΕΦΡΑΓ και ακούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που βοήθησε και στην έγκριση των διεθνών αυτών λογιστικών προτύπων. Τώρα, ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε ονομάζεται Primary Financial Statements. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για τους επενδυτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να προσφέρουμε ε, καλύτερη δομή όσον αφορά τα έσοδα. Γιατί ορίζουμε τα έσοδα απάνω και τις απώλειες κάτω, αλλά ανάμεσα δεν υπάρχουν πολλά. Και όλοι θέλουν να ξέρουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ποια είναι τα υποσύνολα να τα εξετάσουμε για να καταλάβουμε έτσι την απόδοση μιας επιχείρησης. Δεν το κάναμε. Και γι' αυτό υπήρχαν πολλά ε, μέτρα τα οποία υιοθετούσαν τελικά οι ίδιες επιχειρήσεις χωρίς πειθαρχία τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτά τα μέτρα βέβαια πάντα ε, κατέληγαν σε μια καλή εικόνα χωρίς να αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης. Γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε ότι θα ήταν σημαντικό να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι. Αποφασίσαμε λοιπόν να ορίσουμε υποσύνολα και να ζητήσουμε περισσότερη πειθαρχία όσον αφορά τα μέτρα τα οποία δεν προέρχονταν από εμά. Και μάλιστα, επειδή υπήρχε και η ψηφιακή διάσταση χρήσης των στοιχείων. Υπήρχαν όλο και περισσότερα δεδομένα ε, στη διάθεση του κόσμου, και γι' αυτό η πληροφορία πρέπει να είναι διαρθρωμένη και δεν ήταν αρκετά. Ή, αν έχω πρόεδρε ακόμα λίγο χρόνο, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω και για τον ρόλο μας στην ευρύτερη, στο ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς από τις επιχειρήσεις για το οποίο πολλοί μιλούν. Εννοείται ότι μας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα χρηματοοικονομικά πρότυπα και πώς ε, γίνεται η αναφορά από τους διάφορους παράγοντες βάσει αυτών των προτύπων για να ξέρουμε το business model, το επιχειρηματικό μοντέλο δηλαδή ή άλλα στοιχεία, ας πούμε πώς λειτουργεί το δίκτυο της επιχείρησής σας. Τέτοιου είδους πληροφορίες δεν μπορεί κανείς να τις πάρει από τον ισολογισμό ή από τα στοιχεία ε, μιας επιχείρησης γενικά. Όμως ενδιαφέρει τους επενδυτές και γι' αυτό οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να τα συμπεριλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους. Εξού και έχουμε κάποιες μη υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθούμε τις επιχειρήσεις στην κατάρτιση της ετήσιας εκθεσή τους. Επίσης, οι πληροφορίες για τη βιωσιμότητα ενδιαφέρουν και οικονομικά τις επιχειρήσεις. Οπότε ενημερώνουμε αυτή ε, τη δήλωση στα σχόλια λέγοντας στις επιχειρήσεις ότι αν υπάρχουν θέματα βιωσιμότητας τα οποία επηρεάζουν τα οικονομικά σας δεδομένα, όχι απαραίτητα τώρα, αλλά ίσως και στο μέλλον, θα πρέπει να τα συμπεριλαμβάνετε στα διαχειριστικά σχόλια. Είναι ένα μέσο, δεν είναι ότι φτιάχνουμε εμείς πρότυπα βιωσιμότητας, απλώς βοηθούμε τις επιχειρήσεις να μπορούν να τα αναφέρουν. Τέλος, να σας πω και δύο λόγια για το IBOR, γιατί ξέρω ότι πολλοί ανησυχούν στην Ευρώπη. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια ε, όσον αφορά τα επιτόκια και έχουν ε, προκύψει πολλά ζητήματα. Να ξέρετε ότι δουλεύουμε σκληρά, ε, είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να είμαστε έτοιμη ε, έγκαιρα και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι να τα εγκρίνει. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στις ερωταπαντήσεις. Πέντε λεπτά έχουμε εκ μέρους του ΕΛΚ την κυρία Σύρπα Πιτικάινεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Ήθελα να αναφέρω δύο θέματα και να τα τονίσω. Υπάρχει πάντοτε αυτά τα ε, προβλήματα που έχουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες ε, για την κερδοφορία της ρευστότητας. Επίσης υπάρχουν κάποια ζητήματα με τις επενδύσεις ε, όσον αφορά στα ορυκτά καύσιμα που αυξάνουν τους κινδύνους. Επίσης, Υπάρχει και ένας περιορισμός που δεν είναι ηθελημένος από τον κανόνα υπολογισμού των ε, ε, διεθνών προτύπων ε, που έχει να κάνει με τις επενδύσεις και τον κίνδυνο των επενδύσεων. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω από εσάς πώς προτίθεστε να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα και αν έχετε σκεφτεί να κάνετε κάποιες προσαρμογές στον ε, υπολογισμό ε, των LDI, δηλαδή στην λογιστική της βιωσιμότητας, ε, γιατί ούτε εκεί βλέπω ένα εναρμονισμένο σύστημα. Πώς μετράμε και εκεί. Καλό θα ήταν να έχουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στα οικονομικά. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή ε, και με το κλίμα και με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Καλό θα ήταν ε, λοιπόν ε, τα επόμενα χρόνια να υπάρχει και μια εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή ερώτηση και τη λαμβάνουμε όλο και περισσότερο. Ας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει πολύ αυστηρή νομοθεσία για την βιομηχανία πετρελαίου και αερίου. Έτσι θα τους αναγκάσουμε να σταματήσουν πολλές δραστηριότητες ε, εξόριξης τα επόμενα χρόνια. Οι λογιστικές απαιτήσεις ήδη βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που αν υπάρχουν επενδύσεις σε υποδομές, τις επενδύσεις αυτές δεν μπορείς να τις ε, ε, ξανακερδίσεις στην ουσία πρέπει να υπάρχει μία απόσβεση της επένδυσης και να φαίνεται στον ιστολογισμό και στην δήλωση εσόδων-εξόδων. Αυτά ε, είναι πράγματα ε, που ε, θα ισχύουν στο άμεσο μέλλον, τα επόμενα 3-5 χρόνια. Η κανονική λοιπόν λογιστική κάνει τη δουλειά της, δεν χρειάζεται να αλλάξουν πολλά. Υπάρχουν όμως άλλοι κίνδυνοι που είναι πιο μακροπρόθεσμοι. Ε, οι πετρελαϊκές εταιρείες ε, και οι εταιρείες αερίου κάνουν επενδύσεις σε βάθος 10, 20, 30 ετών. Ε, δεν φαίνεται ότι απειλούνται οι επενδύσεις τους γιατί φαίνεται ότι σε αυτό το διάστημα θα κατανελώνεται το πετρέλαιο. Κοιτάνε βέβαια το πολιτικό κλίμα και βλέπουν ότι στο μέλλον θα έχουν πιο αυστηρή ε, νομοθεσία με πιο έτσι ήπιη πληροφόρηση ε, λέγοντας τους ότι αυτά είναι πιο πολύ προς το μέλλον θα μπορούσαμε να ε, βάλουμε κάποιες πρώτες βάσεις ε, και να ε, εξηγήσουμε τι ακριβώς ε, χρηματοοικονομικά μπορεί να συμβαίνει αυτό σε επίπεδο απειλής για την εταιρεία τους στο μέλλον. Έχετε χρόνο για μία επερώτηση, γρήγορη αν επιθυμείτε. Ναι, όντως υπάρχει χώρος για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ήθελα όμως να δω πέρα από αυτά τα ποιοτικά δεδομένα, θα ήθελα και πιο αυστηρούς λογιστικούς κανόνες που να φαίνεται η τόνη, τα γαλόνια, ε, πώς αυτά μεταφράζονται σε επίπεδο επίπτωση στην βιοπικιλότητα από την πλευρά των εταιριών αυτών. Και νομίζω ότι το IFRS ακριβώς ε, ε, αυτό μπορεί να το πετύχει. Είναι ε, πιο ευρία η εφαρμογή του. Γι' αυτό. Ναι, υπάρχουν ήδη πρότυπα και πλαίσια που χρησιμοποιούνται. Ας πούμε, το πλαίσιο της Task Force ε, για τις ε, δηλώσεις περί ε, από το Financial Stability Board. Αυτό κοιτάει πιο μακροπρόθεσμα, ζητά από τις εταιρείες να έχουν μακρόπνα σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η, συζή... η... η κατάσταση. Έχει και ποσοτικά στοιχεία, βέβαια είναι λίγο πιο ασαφή σε σχέση με την λογιστική που κοιτάει στο παρελθόν και καταγράφει αυτό που έχει ήδη συμβεί και είναι πιο αυστηρή. Όμως τέτοια στοιχεία, τέτοιες πληροφορίες σίγουρα έχουν θέση ε, σε ένα management commentary, σε ένα σχόλιο και ε, φυσικά ε, δεν είναι μόνο λόγια, είναι και αριθμοί. Ευχαριστώ εκ μέλους του ISND ο κύριος Λαούμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω έμπειρους ειδικού εδώ στην Επιτροπή μα. Έχω δύο ερωτήσει. Πρώτον, για το IFRS 17 και δεύτερον για το τομέα των ελεγκτών. Είπατε, κύριε Λικάνεν, ότι έχουμε τη διαφάνεια που βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος όταν εξετάζουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον ασφαλιστικό τομέα. Ωστόσο, σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν εφαρμόζουν όλες οι χώρες το πρότυπο 17 και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι οι ΙΠΑ ίδιες δεν το εφαρμόζουν εφόσον ε, εκεί δημιουργήθηκε αρχικά το σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη γνώμη σας, ε, κύριε Λίκαν, που ήσασταν τόσο ενεργός πριν από 18-20 χρόνια. Γιατί και πώς οι δεν το εφαρμόζουν και πώς αυτό επηρεάζει τη διαλειτουργικότητα. Και έπειτα για τον κύριο Χόγκερμποστ έχω μια ερώτηση που αφορά το ρόλο του ε, τομέα ελέγχου. Ε, λογιστικού ελέγχου, γιατί ξέρουμε πως ε, οι λογιστικοί έλεγχοι παίζουν σημαντικό ρόλο εδώ ε, για να δούμε αν όντως λένε την αλήθεια οι εταιρείε για τα οικονομικά τους. Τα πρόσφατα χρόνια είχαμε πολλά σκάνδαλα όπου οι λογιστές έπαιξαν αρνητικό ρόλο. Θέλω να ξέρω λοιπόν ποια είναι η δική σας γνώμη όσον αφορά τη Βρετανία την πρόταση της Βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού για διαχωρισμό των ελεκτικών από τις συμβουλευτικές δραστηριότητες, ώστε να μπορέσουν και εταιρείε εκτός των μεγάλων τεσσάρων να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που χρειάζεται ώστε να μπορούν να προβαίνουν στους ε, ελέγχους ανεξάρτητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πρώην Υπουργό Οικονομίας ε, ο κύριος Χόγκερ Φώστα. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Οι ΙΠΑ αναμίχθηκαν εντόνως ε, στην αρχή και πίεσαν. όμω στη διάρκεια της ε, χρηματοπιστωτική κρίση τα, οι δρόμοι μας χώρισαν. Όμω θέλω να τονίσω ότι οι σχέσει εργασία μα είναι εντάξει και βεβαίω όσον αφορά τι χρηματοπιστωτικέ μας εκθέσεις γίνονται δεκτές στις αμερικανικές αγορές και ε, οι δύο πλευρέ ωστόσο πιστεύουν πως είναι σημαντικό να αποφευθεί οποιαδήποτε ε, πιθανή ρήξη. Όταν δηλαδή υπάρχουν εντάσεις σε διεθνές επίπεδο ε, προσπαθούμε να ε, δισταθούμε. Εγώ ας πούμε πρόσφατα είχα μια συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τους ομολόγους μας. Ε, επισκεφθήκαμε το ICC που είναι η ε, αρχή στον τομέα μας, ε, στη είπα. Επίσης με την ISB συνεργαστήκαμε. Τέλος πάντων, ε, λειτουργούν τα πράγματα. Δεν είναι το ιδανικό, δεν είναι το τέλειο. Θα θέλαμε να έχουμε ακριβώς τα ίδια πρότυπα, αλλά δεν είμαστε ακριβώς τα ίδια. Σε κρίσιμους τομεί ε, έχουμε τα κοινά πρότυπα και έχουμε δεσμευτεί να μην δημιουργούμε προβλήματα. Βέβαια, ταυτόχρονα η διάδοση των δικών μας προτύπων, των διεθνών μας προτύπων, αλλάζει το σκηνικό. Επισκέφθηκα την Κίνα και την Ινδία πρόσφατα και, και την Ιαπωνία λίγο πριν για να δω πώς εφαρμόζεται το IFRS στον κόσμο. Είναι όντως παγκόσμιο πρότυπο πλέον. Περισσότερες εταιρείες το χρησιμοποιούν. Για μας βεβαίως είναι πιο Ε, απλό εφόσον έχουμε την ίδια εφαρμογή σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλύτερο ήταν, θα ήταν βέβαια να έχουμε ακριβώς τα ίδια πρότυπα και με την ΣΥΠΑ, αλλά εφόσον αυτό δεν γίνεται, η αρχή της μη ρήξης και αυτή η ειρηνική φιλική συνύπαρξη λειτουργεί για μας. Εμείς προσπαθούμε να δουλεύουμε διαρκώς ε, για τα διεθνή πρότυπα, ώστε να αποφεύγονται οι διαφορές. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Να πω και εγώ κάτι. Η Αμερική αποφάσισε το 2011 να κάνει και πάλι την Αμερική σπουδαία. Αυτό πολύ μας απογοήτευσε τότε και πολύ προβλέψαμε ότι ο υπόλοιπο κόσμος θα απομακρυνόταν από το EFRS ε ε, τότε. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη τα διεθνή πρότυπα και η χρήση του συνέχισε να αυξάνεται. Πάνω από το 1, πάνω από το 1 τρίτο οι Ιαπωνικών εταιριών χρησιμοποιούν καθαρά, ξεκάθαρο το IFRS και για τα κινέζικα πρότυπα οι διαφορές είναι σχεδόν ε, μηδαμινές και η Ινδία συγκλίνει με γοργούς ρυθμούς. Η σύγκληση λοιπόν από τον υπόλοιπο κόσμο είναι πολύ μεγάλη. Είναι πραγματικά παγκόσμια διεθνή πρότυπα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε παντού. Ελπίζω πως εάν καταφέρουμε να παγιώσουμε τη χρήση του ΕΦΡΕΣ σε όλες τις χώρες και δεν διαλυθούν για να πάνε ο ένας δεξιά και ο αριστερά, τότε και αμερικανικές εταιρείε θα πούν μα καλύτερα είναι να έχουμε και εμεί τα ωφέλη που έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείε που ακολουθούν τα διεθνή ε, πρότυπα και θα το ζητήσουν από μόνοι τους. Τώρα, έχω και προσωπικές απόψεις γι' αυτό. Καταρχάς, η ιδέα όσον αφορά τους κοινού ελέγχους. Είναι καταστροφικό αυτό, γιατί αν δυο ελεγκτικέ εταιρείε καταστούν υπεύθυνε για την ίδια δουλειά, τότε η ατομική ευθύνη διαχέεται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και έπειτα είναι παράξενο όταν πούμε, ναι, ναι, ωραία, οι ελεγκτικές εταιρείε πέτυχαν, οπότε τι να κάνουμε, να διπλασιάσουμε τον το τζίρο τους. Γιατί αυτό θα συμβεί, θα έχουν περισσότερη δουλειά. Και δεν βοηθάει αυτό. Και τέλος, αυτό ενισχύει τις τάσεις του ολιγοπολίου στο, στις λογιστικές εταιρείες και στους ελέγχους, γιατί είναι λίγες οι εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι κακό, λάθος. Νομίζω πως το Ηνωμένο ε, Βασίλειο θα το, το εγκαταλείψει αυτή την ιδέα και να υπάρχει σαφέστερος διαχωρισμός ανάμεσα στις συμβουλευτικές λειτουργίες και τους ελέγχους είναι πολύ καλύτερη ιδέα. Επειδή είμαι επικεφαλής των Επιτροπών Ελέγχου, ε, να σας πω ότι είναι πρόβλημα να έχουμε υποψηφίους για να κάνουν αποκλειστικά και μόνο έλεγχο από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί οι εταιρείε θέλουν να κάνουν και συμβουλευτική δουλειά και αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δεν έχω κανέναν εξ του Ρενιού. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο? Όχι. Και δεν έχω και κανέναν ε, που να θέλει να πάρει το λόγο από το ID. Ο Σβέν Κίγκολτ από τους πράσινους τώρα λοιπόν. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε ενδιαφέρουσε ανταλλαγές απόψεων στο παρελθόν. Τώρα υπάρχουν νέοι ευρωβουλευτέ εδώ. Χαίρομαι που βλέπω και τον κύριο Λίκανεν εδώ, υπό τη νέα του ιδιότητα. Θα ήθελα βέβαια και άλλες προτάσεις σας να γίνονταν αποδεκτές από τους νομοθέτες όσον αφορά για παράδειγμα τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των τραπεζών. Τώρα είναι ενδιαφέρον που σας βλέπουμε από αυτήν την ιδιότητα. Θέλω να υποφεληθώ επίσης από την ευκαιρία αυτή για να προσπαθήσω να δω λιγάκι το θέμα της συνεργασίας μας. Άκουσα τι είπατε. Και εννοείται ότι το μεγάλο σχέδιο αυτή και το μεγάλο πρόγραμμα τη θητεία αυτή είναι η Πράσινη Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει ότι στηρίζει ευρέω την Πράσινη αυτή Συμφωνία και συζητιέται το θέμα των λογιστικών προτύπων. Τι σημαίνει δηλαδή αυτή η συμφωνία για τα λογιστικά πρότυπα. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Χόχερ Φόρστερ να λέει ότι είναι εντάξει και διαβάσαμε και το έγγραφο του κύριου Άντερσον που λέει ουσιαστικά ότι θα δούμε πώς θα επιβαρυνθούν οι δηλώσεις, οι χρηματοοικονομικές εν καιρό. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν φτάνει. Και δεν είναι αυτό το οποίο ε, περιμένει ο κόσμος και οι ενδιαφερόμενοι από εσά. Είναι λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για σας τώρα, Όπω και στο παρελθόν, όταν μιλούσαμε για τα φορολογικά ζητήματα. Τώρα έχουμε το IASB, τον Οργανισμό δηλαδή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και πρέπει εσείς να πείτε αυτό ζητάμε. Και το πώς θα αντιδράσετε εσείς ε, θα μας δείξει και κατά πόσο ανταποκρίνεστε ή όχι στις προσδοκίες μας. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες χώρες έχουν εκπροσώπους δημοκρατικά εκλεγμένους και ο δικός σας οργανισμός θα πρέπει να είμαστε ξέρουμε ότι δεν συνδέεται με το θέμα αυτό των εκλογών, των δημοκρατικών εκλογών και ίσως η Ευρώπη θα έπρεπε να το ξαναδεί αυτό από πλευράς αρχής. Απάντηση Λίκανεν. Για το δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει σύνταγμα, έτσι. Τι έχει αλλάξει. Όσον αφορά τη δικιά μας τη δομή, έχουμε το δικό μας ελεγκτικό συμβούλιο, την Επιτροπή και υπάρχουν και οι τραστείς που είναι πιο κάτω. Καταλαβαίνω όμως τι λέτε και εντάξει θα μας προβληματίσει ως δυνατότητα. Δεν είναι απλό όταν ένας οργανισμός είναι παγκόσμιος και έχει 140 χώρες, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε εκλογέ όπως λέτε, αλλά πάση περιπτώσει είναι κάτι που συνεχίζουμε να το συζητάμε. Τώρα ένα σχόλιο για την Πράσινη Συμφωνία. Εννοείται ότι παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη διάβασα. Υπάρχει ο Κρίστιαν Γκολφιέρ, Γάλλος οικονομολόγος, που έβγαλε ένα βιβλίο το Φεβρουάριο και είπε ότι το πιο ενδιαφέρον είναι ο φόρος επί του άνθρακα. Όμως αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουν με το στόχο που είναι καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και προτινόμενα μέτρα για να το πετύχουμε αυτό. Άρα πρέπει ο πολιτικός κόσμος να συμφωνήσει και αυτό είναι το περίπλοκο. Πάντως γενικά, εννοείται ότι στο IFRS Θέλουμε να βοηθήσουμε τους επενδυτές και παρακολουθούμε τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλουμε να συμβουλεύουμε τους επενδυτές, οι οποίοι λένε ότι έτσι κι αλλιώς εμείς ένα νούμερο θέλουμε να μας δίνετε. Και τελείωσε. Ναι, αλλά δεν φτάνει. Τι άλλο συμβαίνει εκεί γύρω. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τελικά για τους επενδυτές ε, πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν καλύτερα για τις επενδύσεις τους και η Πράσινη Συμφωνία είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Θα επανέλθουμε πάντως και ευχαρίστω να το ξανασύστησουμε και αργότερα. Χόχερφόρστ. Δεν θέλω να πω ότι όλα είναι τέλειο όσον αφορά τη βιωσιμότητα κλπ. Όχι, δεν είναι αυτή η εικόνα που θέλω να δώσω και στις ομιλίες μου το λέω ότι λυπάμαι που είναι τόσο πολλοί παίκτες και υπάρχει τέτοιο κατακαιρματισμό στο θέμα της βιωσιμότητα. Κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ. Ότι είναι δύσκολο, ναι. Τι ρόλο εμείς μπορούμε να παίξουμε, ούτε και αυτό είναι ξεκάθαρο ακόμα για μας. Σκεφτόμαστε πάντως. Και υπάρχουν δύο ειδών ε, πρότυπα βιωσιμότητα. Το ένα που συνήθω κοιτάμε είναι τα θέματα βιωσιμότητας για το οικονομικό μέλλον μιας επιχείρησης. Αλλά υπάρχουν και άλλα πρότυπα βιωσιμότητα εξίσου θεμητά, αλλά πολύ διαφορετικά, που είναι να ρωτήσουμε την επιχείρηση εσείς τι κάνετε για τον πλανήτη, τι κάνετε για την κοινωνική σταθερότητα, για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι βέβαια στο δικό μας DNA, μπορούμε να το μελετήσουμε όμως, να το επεξεργαστούμε τα άλλα τα πρότυπα που σας ανέφερα πριν ανταποκρίνονται καλύτερα στην εντολή μας και την αποστολή μας. Αλλά τα σκεφτόμαστε και αυτά. Και σίγουρα εγώ δεν θέλω να υπονοήσω ότι όλα είναι τέλεια. Όχι. Αλλά να πω ότι αν το θέμα είναι σοβαρό για μια επιχείρηση, θα βρει τον τρόπο να το αντικατοπτρίσει και στην οικονομική της πολιτική. Ο κύριος Έπινγκ από το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι για την παρουσία εδώ και των δύο. του γνωρίζω και του δύο, τον κύριο Φόρστο για αρκετό καιρό, τον κύριο Λικάνεν από τότε που ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δούλευα και εγώ τότε στον κύριο Χόγκενστάιν. Ο κύριος Ρέν ήταν επικεφαλής του γραφείου του. Λοιπόν, Αγαπητοί κύριοι, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπέρ τη πράσινη συμφωνία που αναφέρθηκε για να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δαπανίσει δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια, σε πράσινα προγράμματα και η ΕΚΤΕ σκοπεύει να εκδώσει κοινά πράσινα ομόλογα. Όμω δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι επενδυτικά προγράμματα είναι πράσινα και ποια δεν είναι. Η πιστοποίηση λοιπόν πρέπει ακόμα να αποφασιστεί. Οπότε ρωτάω, εσείς όντας ε, το οργανισμός ε, προτύπων, λογιστικών προτύπων, εσείς πώς ε, καταλήγετε στο ότι είναι πράσινο και τι δεν είναι. Δεν υπάρχει κίνδυνος πολιτικής καθοδήγησης τελικά. Η πράσινη συμφωνία μπορεί τελικά να αφαιρέσει τον ανταγωνισμό από την εξίσωση και να καταλήξουμε σε ένα σύστημα επιδοτήσεων κρατικών που πληρώνονται τελικά από τον φορολογούμενο. Οπότε τελικά καταλήγουμε σε μια ε, οικονομία που σχεδιάζεται κρατικά. Μα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το πρόβλημα, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Χόχερφόστ. Η ζωή πρόεδρος του IASB είναι αρκετά περίπλοκη ως έχει ε, έχει μέσα και λίγη πολιτική, ακόμα και τα λογιστικά πρότυπα έχουν μέσα λίγη πολιτική και πολύ χαίρομαι που δεν είμαι εγώ που καλούμε να λύσω αυτά τα προβλήματα. Είναι εκτός δικιά μου εντολής, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι η δημιουργία μιας πράσινης ταξινόμησης είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Διάβασα σε εφημερίδες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αφήσει την πυρηνική ενέργεια εκτός ε, του πράσινου κομματιού. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το σκεφτεί κανείς αυτό. Οπότε είναι πολιτική τελικά η απόφαση για το αν είναι ή δεν είναι κάτι πράσινο η πυρηνική. Αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή, έτσι. Οι πολίτες το σκέφτονται, το συζητάνε, αλλά δεν θα ήταν σοφό εγώ που είμαι πρόεδρος του ISB τώρα να πω Πρώτα απ' όλα δεν έχω καταλήξει καν εγώ ίδιος. Οπότε πώς να καταλήξω εγώ σε λύση ενός τέτοιου προβλήματος. Και ο κύριος Λικάνεν, δύο σχόλια έχω να κάνω για τον ε, φόρο στον Ανθρακά. Η Φιλανδία ήταν η πρώτη χώρα που πρότεινε να υιοθετηθεί ένας τέτοιος φόρος, που δεν ήταν βέβαια δημοφιλής, αλλά εφαρμόστηκε και μας ακολούθησε και η Σουηδία στη συνέχεια. Η βασική λογική λοιπόν της οικονομίας τι είναι. Είναι αν οι εξωτερικεύσεις ε, δουλέψουν καλά, μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Και όταν φτάνουμε σε αυτή την πράσινη χρηματοδότηση, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι εννοούμε. Να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και ταξινόμηση αυτή η πράσινη που θέλουμε να κάνουμε σε επενδύσεις είναι κάτι σημαντικό. Εγώ προσπάθησα να διαβάσω ολόκληρο το έγγραφο, δεν είναι βέβαια κάτι εύκολο να καταλάβει και μαθαίνουμε βέβαια όσο περνάει ο καιρό και μπορεί κάλλιστα να γίνει πιο ξεκάθαρο το έγγραφο για να αποφύγουμε και το περίφημο greenwashing, δηλαδή να παρουσιάζονται σαν πράσιμες επενδύσει κάποιε που δεν είναι, να είναι μόνο σε επίφαση. Είναι πάντως κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο και θα δούμε τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε εμείς. Ε, παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα πάντως, να ξέρετε. Ευχαριστώ. Δεν έχω κάποιον άλλον από την ΚΟΕ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος δεύτερος ε, που θέλει να λάβει το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ. Όχι, τότε δίνουμε τον λόγο στους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Τάγκ. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζω τη σημασία της συζήτησης για το IFRS 17 και για τον ασφαλιστικό τομέα, αλλά εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε ένα άλλο θέμα, πιο στρατηγικό. Με έχει λίγο μπερδέψει η παρουσίαση, γιατί μιλάτε πάρα πολλές φορές για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας, αλλά όταν μιλάω για ένα Γάλλο, με έναν Γάλλο ή Γερμανό διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων ζητούν απεγνωσμένα δεδομένα, ε, περισσότερα δεδομένα. Δεν τους ενδιαφέρει η βιωσιμότητα γενικότερα. Ε, για την ίδια τη βιωσιμότητα της εταιρεία του σε κρηματοοικονομικό επίπεδο παλεύουν και πασχίζουν. Ε, γι' αυτό ζητούν ε, όλο και περισσότερα δεδομένα και προσπαθούν να τα βρουν με κάποιο τρόπο. Είπατε λοιπόν ότι το συζητούσατε αυτό. Όμως δεν είναι και προφανές δεν απορρέει προφανώς από όλο αυτό ότι πρέπει να τυποποιηθούν και πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα δεδομένα των εταιριών, με την ταξινομία και μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων, ε, ίσως προς αυτή την κατεύθυνση να πιέζουμε τελικά. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, ξέρω και είναι δεδομένο όπως το ξέρετε κι εσείς, ότι οι θεσμικοί επενδυτές ε, της Ολλανδίας ε, που έχουν κάνει τον ε, σύνδεσμο γεωμήλων θέλουν πάρα πολύ τέτοιες πληροφορίες. Και μάλιστα έχουν στείλει και ένα έγγραφο και μας ζητούν να το κάνουμε εμείς αυτό. Το εξετάζουμε. Οι τραστείς αυτή τη στιγμή εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο. Να σας πω όμως το εξής. Όποιες και είναι οι περιστάσεις αυτό που είναι πιο σημαντικό για μας ε, είναι το σημερινό μας ε, πεδίο εντολής. Ε, δεν είναι βέβαια επαπειλούμενο. Η βιωσιμότητα είναι ένα κομμάτι Τώρα εμείς βέβαια ασχολούμαστε περισσότερα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα λογιστικά δηλαδή στοιχεία. Στο παρελθόν όταν έγινε εγώ πρόεδρος κανείς δεν ασχολείται με την βιωσιμότητα. Τώρα στο Management Commentary έχουμε δημιουργήσει χώρο για την βιωσιμότητα. Άρα ε, προβλέπουμε, κάτι κάνουμε. Τώρα ο βαθμός στον οποίο μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Φυσικά μπορούμε να προστατευτούμε στους σύγχρονους καιρούς, αλλά πάντοτε πρέπει να προσέχουμε να μην μπαίνουμε σε χωράφια που δεν είναι στο DNA μας. Αυτό λοιπόν είναι και το ερώτημα που μας ταλανίζει αυτή τη στιγμή. Το του λεχθέτος ε, βλέπω ότι υπάρχει ανάγκη για σωστή ε, αναφορά και πληροφόρηση σχετικά με τη βιωσιμότητα είναι πιο δύσκολο, δεν είναι ε, χρηματοοικονομική αναφορά με τη μορφή που ξέρουμε ως τώρα, ε, κοιτάει προς το μέλλον, είναι λιγότερο ακριβής ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Και καταλαβαίνετε, η λογιστική ήδη έχει πολλές πολιτικές διαστάσεις, θα γίνει ακόμα πιο μεγάλο το πολιτικό βάρος ε, σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο λοιπόν το ερώτημα για να το απαντήσω και είμαστε πολύ προσεκτικοί. Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι το σκεφτόμαστε. Θέλετε περώτηση ή μια γρήγορη περώτηση. Ελπίζω ε, και η χρηματοοικονομική πληροφόρηση να κοιτάζει προς το μέλλον. Ε, αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική, είναι κρίσιμη. Δεν περιμένω λοιπόν από εσά να έχετε μια ε, συνολική, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Απλώς με ανησυχεί ότι αν συνεχίσετε να μιλάτε και δεν αρχίσετε κάποια στιγμή, ε, γιατί υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν, Κάποιος όμως πρέπει να ξεκινήσει για να αρχίσει να αναπτύσσει κάτι. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν ήδη πολλά σώματα, πολλοί οργανισμοί στον κόσμο που αυτό το κάνουν ήδη. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά το GRI, το SESB, είναι εκεί ήδη και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Εγώ θα ήθελα πραγματικά όλοι αυτοί να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, ίσως και να συγχωνευτούν και να δημιουργήσουν έναν τομέα παγκοσμίων προτύπων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του, αλλά γενικά καλό θα ήταν να έχουμε παγκόσμια πρότυπα για αυτό το πρόβλημα. Γιατί όπως είπατε είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο πρόβλημα με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εγώ μιλώ με όλους και ο Έρκη μιλάει με πολύ κόσμο. Το σκεφτόμαστε λοιπόν. Αλλά αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με μεγάλη προσοχή. Ωραία. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα για όποιον θέλει στην διαδικασία Κατστιάη να λάβει το λόγο. Ο κύριος Γιακελούνιας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Λικάνεν, ε, πραγματικά η διαφάνεια που δείξατε με το χάσμα μεταξύ των αποδόσεων επενδύσεων ε, και το τι συμβαίνει στην Γερμανία και στην ε, Ιαπωνία αντίστοιχα με έβαλε σε σκέψεις. Είναι ένα πολύ δύσκολο και περίπλοκο θέμα σε επίπεδο λογιστικής, αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς των καταναλωτών. Γνωρίζετε για πόσο καιρό αυτές οι προβολές, αυτές οι προβλέψεις των πραγματικών επιτοκίνων θα μπαίνουν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών γιατί υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι αυτό μπορεί τα αρνητικά πιστόκια δηλαδή να συνεχίσουν για δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις εταιρείες αυτές, ε, κάποιοι όμιλοι μπορεί ε, να ε, μην μπορέσουν να ορθοποδήσουν αν συνεχίσει αυτό το προεξοφλητικό επιτόκιο να είναι αρνητικό συνεχώς. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Κάποιες ε, χώρες όπως η Κορέα έχουν μεγάλο θάρρος. Η, η Κορέα θα εγκρίνει, θα υιοθετήσει το IFRS 17 και θα προσπαθήσει να κεφαλοποιήσει αυτό το θέμα σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιριών, γιατί πραγματικά ε, εκεί χρειάζονται πολλά κεφάλαια οι ασφαλιστικές σε αυτό το θέμα πολλοί Γερμανοί ασφαλιστές ε, που είναι εκτός του πεδίου του IFRS, είναι μικρές, μικρότερες εταιρείες, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και τι να πω, ελπίζω και η Ευρώπη κάποια στιγμή να επιταχύνει τη διαδικασία επικύρωσης. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο καλύτερα θα συνεχίσουμε για πολύ καιρό. Εγώ είμαι Ήμουν σε μία χώρα όπου οι ντόπιοι ασφαλιστές μου είπαν ότι ο, η ρυθμιστική αρχή δεν τους επιτρέπει να προσφέρουν κάποια συγκεκριμένα προϊόντα γιατί ε, οδηγούν σε ζημίες και πρέπει να πάνε σε εναλλακτικά προϊόντα. Γενικά, καλό είναι να είμαστε σίγουροι για το τι θα συμβεί και τα πράγματα δεν φαίνονται ακόμα πώς θα εξελιχθούν. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο πιο εύκολα θα προβλέψουμε τα προβλήματα και γιατί πραγματικά το θέμα είναι πολύ μεγάλο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ακόμα και οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι κάτω από τη λογιστική αξία και αυτό για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Σε μια ήπειρο που πολλές τράπεζες είναι ακόμα ασθενείς, το πρόβλημα γίνεται πολύ σοβαρό. So no more... Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά το λόγο. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Χόχερφος και τον κύριο Λικάνε. υπάρχει άλλο ένα κατσδιάι και έχουμε χρόνο. Παρακαλώ. Merci de me donner la parole. Moi, je revenais sur... Alors, je... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι και εκ νέου σε αυτή την επιτροπή. Ε, είμαι δηλαδή νεοφερμένος και δεν ε, ξέρω ακριβώς τι γίνεται με το περιεχόμενο των κανόνων ε, βιωσιμότητες. Σε κάποιες χώρες έχουμε υιοθετήσει τις αναφορές ε, που είναι υποχρεωτικές για τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αυτές ενδιαφέρονται και για τα διεθνή πρότυπα, όπως τα λένε, ε, καθολικά πρότυπα, που σημαίνει την θετική και αρνητική παραγωγή των εταιριών στην επικράτειά τους. Οι εξωτερικεύσεις ε, ε, σχετίζονται με τη βιοπικιλότητα, δημιουργία δηλαδή θετική, την ευημερία στην επικράτεια, δηλαδή εκεί πρέπει να βρούμε δείκτες για να το μετρήσουμε, αλλά γίνονται σχετικές προσπάθειες και έπειτα η καταγραφή των αρνητικών εξωτερικεύσεων. Μιλήσατε για ισολογισμό διοξιδίου του άνθρακα, αρνητικός αντίκτυπος στη βιοπικιλότητα, ο, οτιδήποτε είδους αντίκτυπο μπορεί να έχει η εταιρεία στην ε, επικράτειά της. Ε, ε, στην περιοχή όπου βρίσκεται. Πιστεύετε πως υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ όμως να είστε σύντομοι. Ξέρω πως στη Γαλλία υπάρχει ε, κανονισμός που ήδη ισχύει και που ζητά από τις εταιρείες να δώσουν πληροφορίες για ένα ευρύτατο φάσμα ε, θεμάτων. Η γαλλική ετήσια έκθεση, ο συλλογισμός είναι πολύ μεγάλος, 400 ε, σελίδες, δηλαδή 50% παραπάνω από ό,τι στη Γερμανία. Και Απαντώντα και στον κύριο Τάγκ που βασικά έθεσε την ίδια ερώτηση με εσά, να καταστήσω σαφές ότι είναι σίγουρο ότι ε, το δικό μα Συμβούλιο θα μείνει εστιασμένο στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δίνουν ε, ε, ε, για, ε, σε ευρύτερο πεδίο και οι τραστείς το κάνουν αυτό με πολύ προσεκτικό και λεπτομερή τρόπο αλλά πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν μπορούμε να επεκτείνουμε και να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Ευχαριστώ τους ομιλητές μας και η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 12. Hello. If everybody can take a... Παρακαλώ, καθίστε. Okay. Before starting the... Ωραία, πριν ξεκινήσουμε τις επίσημες ψηφοφορίες, παρακαλώ να κάνουμε ένα τεστ. Άρχεται η ψηφοφορία, η δοκιμαστική ψηφοφορία. We, think we are... Yes. Είμαστε εντάξει. Άλλοι τρεις απομένουν για να ψηφίσουν. Άλλος ένας. Παρακαλώ να είμαστε σίγουροι ότι όλοι είναι εδώ. Άλλος ένας. Πέρα στις ψηφοφορίες. Okay. So now we can start... Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν και ψηφίζουμε την πρώτη έκθεση ε, για την Τραπεζική Ένωση, ετήσια έκθεση 2009, ε, συμβαστική α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 60, υπέρ, πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ. Ε, να ελέγξουμε. Κάνουμε έλεγχο για την τροπολογία 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική D, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική ή e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 108 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 136 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 126 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 125. Υπέρ. Εκατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ πρέπει να ελέγξουμε. Φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά θέλω να σιγουρευτώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ορίστε. Κάποια χέρια δεν είχαν σηκωθεί από την αρχή. Συμβαστική. Συγγνώμη, παράγραφος 11, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική π, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Q, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AA υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 211 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 236 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ναι, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία να ελέγξουμε τη 237. Πέρας της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 239. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική AB. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 276. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική ΑΕΦ, Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφα 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στα citations, ε, στις αιτιολογικές σκέψεις. Ε, ε, ένα ως τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ, τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, το πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 6. Ε, βλέπω ότι υπάρχει μια προφορική τροπολογία, όχι. Από το Renew. Είμαστε στην 6. Αιτιολογική αναφορά 6. Υπάρχει προφορική τροπολογία από το Renew. Αυτό έχω γράψει. Υπάρχουν ε, κάποιες αντιρρήσεις σε αυτό. Όχι. Υπέρ του oral, του εις προφορικής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην αιτιολογική αναφορά 7 9 unblock. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αρχικό κείμενο, πρωτότυπο κείμενο. Συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε unblock από το 11 ως το 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μία προφορική τροπολογία από τον εισηγητή για την αιτιολογική αναφορά 14. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η έξι καταπίπτει. Άλλη μια προφορική τροπολογία από τον εισηγητή για την 14β. Ε, Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τις τροπολογίες 8 και 9 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε εν μπλοκ. Ε, τιολογικε αναφορες αναφορές 15-22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο αναφορά 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά από αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο αναφορά 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε αν μπλοκ τις αιτιολογικές αναφορές 25-27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική W. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική Y. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική Z. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε στο το κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία όσο έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 42 υπέρ και 9 κατά 3 αποχές. Okay. Now Ωραία, συνεχίζουμε και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της πολιτικής ανταγωνισμού. Ξεκινάμε με την τροπολογία αριθμός 31. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Σ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 241 υπέρ, κατά, Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Εψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική D, δέλτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική G ζήτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική H ήτα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I, Ι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 136, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αν ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Close the vote. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Uh, so 139 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ κατά αποχές. Εδώ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της φοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική L. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική M. Μη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1, νη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 178 υπέρ, κατά, αποχές, εδώ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά. διαφορά. Συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική π. A. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Α, όχι, στην τροπολογία 202 πάμε τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εδώ πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική Q υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 194 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική T τάφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική U υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 239 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 240 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 244 υπέρ, κατά, αποχές, Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. 246 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 112 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 274 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε. 257 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φαίνεται, αλλά ωραία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Γιατί 257 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 263 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 270 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική X υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 119. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική Y, Y υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική αλφα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 298 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. αλφα ΑΣ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε εδώ ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 299 υπέρ, κατά, αποχές, Μπορείτε παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας καλά. Να ελέγξουμε. Ωραία, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 299. Τέλος. Απορρίπτεται. Το υπέθεσα, αλλά πρέπει να σηκώνετε τα χέρια. 301 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 302 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 303 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΓ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 327 τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 329 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑH υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΙ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 335 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 1 στις αιτιολογικές αναφορές υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4, που είναι ίδια με την τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε προφορική τροποποίηση στην αιτιολογική αναφορά 17β. δεν υπάρχουν αντιρρήσει. ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, συμβαστική ΑJ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΚ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, προφορική τροποποίηση στην ελληνική σκέψη C, γ. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 1 της ίντα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάλι ένα δεύτερο τμήμα της ίντα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ίντα 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 5 κατά και 18 αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν. Τώρα, για το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, κανονικά θα ψηφίσαμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο για τον Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής για το 2020. Please. Παρακαλώ ησυχία. Ένα λεπτό σας ζητώ ακόμα για αυτή τη σημαντική ανακοίνωση. Οι συντονιστέ σήμερα το πρωί συμφώνησαν να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου για το θέμα του εξαμήνου, για, ώστε στις 4 Μαρτίου δηλαδή, στις 8.30 το πρωί, να ψηφίσουμε. Περιμένουμε μόνο την έγκριση που θα έχουμε μέχρι το τέλος της απόψινης μέρας. Θα σας το επιβεβαιώσουμε για την ψηφοφορία για αυτή την έκθεση στις 4 Μαρτίου, 8.30 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα συνεδρίασης.